Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο σημείο θα είναι η έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχέση με την Λατινική Αμερική. Τον είδα τον κύριο Σαλαφράγκα. Δεν τον βλέπω όμως τώρα εδώ στην αίθουσα. Τον είχα δει πιο πριν. Πολύ ωραία. Τον είδα να μπαίνει στην, αίθουσα της Ολομέλειας. Ίσως κάποιος από την ε, δική του κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να προσπαθήσει να βρει τον εισηγητή να έρθει στην αίθουσα. Δεν μπορώ να δώσω τον λόγο ούτε στην κυρία Άστον διότι έχει και εκείνη κάτι σημαντικό φαίνεται εκτός Ολομέλειας, εκτός αίθουσας Ολομέλειας. Διακόπτουμε λοιπόν την Ολομέλεια τις εργασίες μας για δύο λεπτά αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόεδρος, εντάξει αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να συνεχίσουμε και θα διακόψει τη συζήτησή του ο κύριος Αλαφράγκα ένα λεπτό και θα πάρει αμέσως τον λόγο. Βρίσκεται καθοδόν τώρα προς τη θέση του. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά για όλους μας. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη συζήτηση για την έκθεση Σαλαφράγκα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε τον λόγο τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Eh, ναι. Κυρία Πρόεδρε, έρχεται η κυρία Άστον, είναι καθοδόν. Θα μπορούσαμε να την περιμένουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να έρθει, για να μπορέσει να ακούσει και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να, τι κατεβαίνει. Δεν το κατάλαβα. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ειδού μπορούμε να έχουμε και το άλλο άτομο στην αίθουσα. Λοιπόν, για τρίτη φορά ξαναξεκινάμε. Λοιπόν, λοιπόν. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε τον λόγο εσείς ως εισηγητής. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπατή Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση, όπω ενεκρίθη από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αφενός αναγνωρίζει την όθηση που έδωσε η Ισπανική Προεδρία που δεν βλέπω εδώ στην αίθουσα, παράγμα που με παραξενεύει διότι συζητούμε για την Λατινική Αμερική και θα ήθελα να καλωσορίσω και την ανακοίνωση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο ε, πολύ μεγάλες ε, περιοχές οι οποίες είναι σε εταιρική σχέση. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα συναντήσουμε άλλες δύο περιοχές που θα έχουν τόσο πολλά κοινά συμφέροντα όπως είναι η Λατινική Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία είναι γνωστά ποσοστά άνω του ενός δις ε, ε, πολιτών και με την Καραϊβική μαζί είναι σχεδόν το 1 τρίτο των χωρών που αποτελούν τα Ηνωμένα Έθνη. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ε, ότι υπάρχει μια μικρή μείωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ακόμα ο μεγαλύτερος δωρητής στις χώρες Λατωνικής Αμερικής και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος. Πέρα όμως των στοιχείων, αυτό που αναγνωρίζουμε ε, είναι ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωση ε, Λατινική Αμερική είναι κάτι παραπάνω από μια αγορά. Υπάρχουν κοινέ αξίες όπως είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών, η ελευθερία έκφρασης, το κράτος δικαίου, ε, και ο σεβασμός ε, των νόμων και η άρνηση οποιασδήποτε μορφής δικτατορίας. Και αυτή η σύνοδος φτάνει σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χρονική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την μεταρρύθμιση και την έναρξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα με την χρηματοοικονομική κρίση. Για πρώτη φορά διαπιστώσαμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρέπει μόνο να βοηθήσει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά μια χώρα μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Όταν βλέπουμε τα ποσοστά ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πέρσι είχαμε αρνητική ανάπτυξη, μείον 0,5% ενώ η Λατινική Αμερική είχε μείον 1,8%. Και όταν βλέπουμε και τα στοιχεία της προγνώσης ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ποσοστό ανάπτυξη τη τάξη του 0,7% και η Λατινική Αμερική 5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επόμενη σύνοδο δεν θα είναι μία σύνοδο βορρά-νότου όπω ήταν στο παρελθόν, αλλά θα είναι μία σύνοδο μεταξύ ίσων. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε και λίγο στο παρελθόν και να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος και ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρία Άστον, από το 2000 έως το 2010 θεωρούμε ότι οι, τε, οι συμφωνίες διασύνδεσης με την ε, Χιλή και την Κεντρική Αμερική, όπως επίσης οι συμφωνίες που είχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε με όλη την Κεντρική Αμερική και πολλές χώρες της Μερκοσούρ, δείχνουν ότι πρέπει να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο, θα πρέπει να αναζητήσουμε ενώσουμε τις ε, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις κατά κάποιο τρόπο με τον ε, Μεξικό και τη Χιλή και να δώσουμε νέα αίθουσα σε αυτές τις συμφωνίες, να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική που θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερε δόσεις γενοδορίας και επίση ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλωσορίσουμε και τι πρωτοβουλίε που παρουσιάσατε εσείς ε, για την δημιουργία της λατινοαμερικανικής Ένωση και Ευρωπαϊκής Ενώσεω, και να υπενθυμίσω ότι η σύνοδος αυτή, κυρία Άστον, δεν θα είναι μία ακόμα σύνοδος. Πρέπει να συζητήσουμε ένα πολύ σαφές ζήτημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε έδαφος στα εμπορικά θέματα με την περιοχή, ε, και να τα χάνουμε και από χώρε όπω είναι η Κίνα, θα γίνουμε πραγματικά άσχετοι για αυτού. Γι' αυτό ακριβώ ε, σα ζητώ, κύριε Άστον, ω είπατε εκπρόσωπο και ω αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αποστείλετε ένα πολύ σαφέ μήναμε για τη δέσμευση τη Ευρώπη που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε και την εταιρική σχέση με του φίλου τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου, κύριο Σαλαφράγκα. Συγγνώμη κύριε Σαλαφράγκα, δεν άκουσα την τελευταία σας παρέμβαση. Είχε κλείσει το μικρόφωνο, δεν άκουσα τα ισπανικά σας. Αλλά θα σας δοθούν δύο λεπτά στο τέλος. Αν ρωτήσατε αυτό, η απάντηση είναι ναι. Τέσσερα λεπτά στην αρχή και δύο στο τέλος. Συγγνώμη, συνεχίζω στα γερμανικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Άστον τώρα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένω τη συζήτηση ε, για τις σχέσεις ε, με τη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα για την εξαιρετική του έκθεση. Νομίζω ότι καταδεικνύει τη σύγκληση απόψεων μεταξύ των δύο ε, θεσμικών οργάνων μας και δείχνει επίσης και τις προοπτικές των εταιρικών σχέσεων που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την περιοχή. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με την Λατινική Αμερική ε, και θεωρούμε ότι μια συντονισμένη προσπάθεια θα σημαίνει ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή. Και η επερχόμενη σύνοδος είναι ένας καλός τρόπος ε, να επανεπισημάνουμε την αποφασιστικότητά μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Και όπως υπόθηκε, ήταν επιτυχής η εταιρική σχέση. Είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος επενδυτής στην περιοχή και θέλουμε να καλύψουμε και άλλους στρατηγικούς τομείς, την κλιματική αλλαγή, τη μη διασπορά των όπλων, την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρσι υπήρξε μία ανακοίνωση, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική είναι παγκόσμιοι εταίροι σε συνεργασία. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε βάσει αυτού την περιφερειακή ολοκλήρωση, να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσει, ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την ποικιλομορφία της περιοχής, να έχουμε προγράμματα στοχευμένα προς το ε, επιθυμητό αποτέλεσμα. Και επίσης βέβαια έχουμε και πολλές πρωτοβουλίες. Συνεργαζόμαστε με το Μεξικό, με τη Βραζιλία για τη στρατηγική εταιρική σχέση και με τη Χιλή ε, για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη. Με την Κολομβία έχουμε ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει μια πολυμερού εμπορική συμφωνία και αναμένουμε ολοκλήρωση ε, ε, συμφωνιών και με την Κεντρική Αμερική ε, στο πλαίσιο τη Μερκοσούρ. Θέλουμε να έχουμε περισσότερο διάλογο για πολλά ζητήματα όπω η μετανάστευση, η καταπολέμηση των ε, ναρκωτικών. Ε, είναι όλα αυτά τα ζητήματα πέραν των οικονομικών θεμάτων που ενισχύουν την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη συνεργασία μας. Ε, είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε τη Λατινική Αμερική να επικεντρωθεί σε βασικά ζητήματα. Για τη Σύνοδο θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με την επιστήμη, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, θα αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει γίνει με πολλέ ε, ε, υποπεριφέρειε, όπω είπε και ο κύριο ε, Σαλαφράνκα. Τρίτον, ενίσχυση του Ταμείου Επένδυση, συγγνώμη, ίδρυση του Ταμείου Επένδυση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική σε έναν ολοένα και μεταβαλλόμενο κόσμο κόσμο και επίση να αξιοποιήσουμε, να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει. Αναμένω εναγωνίω ε, τι απόψεις των Ευρωβουλευτών ε, και με χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσει τους. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Αστον. Τώρα θα λάβει τον λόγο για την παρουσίαση τη γνωμοδότησης τη Επιτροπής ανάπτυξη. η κυρία Γκρέζε. Δύο λεπτά παρακαλώ. Chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από, το σύνοδο της τη Σύνοδο της Μαδρίτης, ε, σε μια κρίση ε, οικονομική και περιβαλλοντική, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ρόλο να διαδραματίσει, ε, να βοηθήσει και επειδή είναι και πρωτοστάτη στην αναπτυξιακή ενίσχυση, την Λατινική Αμερική με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμεί χαιρόμαστε όλου ιδιαίτερω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να σεβαστεί του αναπτυχιακού στόχου τη χιλιετία για την κατάρτιση και την εκπαίδευση και είδα στην έκθεση ότι αναφέρονται και οι γυναίκε και η προτεραιότητα της καταπολέμησης κλιματική αλλαγή. Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα μέτρα, δεν υπάρχουν ε, πραγματικέ στρατηγικέ για την ανάπτυξη. Μετά από την Κοπενχάγη, η Επιτροπή Ανάπτυξη, είχε ζητήσει ε, καινοτόμα προγράμματα στη Λατινική Αμερική, όπω ακούσαμε αυτήν την εβδομάδα, ή όπω τα προγράμματα που είχαμε στον Ισημερινό. Ο σεβασμό των πολιτικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών είναι στο επίκεντρο των ε, ανησυχιών και των ε, ε, πρωτοβουλειών μας. Αν δεχθούμε την κατάσταση στην Κολομβία, ε, δεν ε, θα οδηγηθούμε σε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να, να γίνουν σεβαστέ οι διάφορε προδιαγραφέ. Ε, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει τη θέση του σε μια έκθεση Επιτροπή Εξωτερικών. Επίση, δεν πιστεύω ότι πρέπει να πολλαπλασιάζονται τα διάφορα προγράμματα με ελάχιστους προπολογισμού που δεν δίνουν τη δυνατότητα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Δεν συμφωνώ με περισσότερες γραμμέ προπολογισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια, για, για αμφί, γιατί η η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξη. Η Λατινική Αμερική δεν είναι ο μόνος αποδέκτης. Έχουμε το Περού, έχουμε και την Κολομβία ε, και αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αντιπαράδειγμα. Ε, θέλουν, δεν, δεν πρέπει να υπάρξει συμφωνία που αποδυναμώνει ε, τα κεκτημένα μας. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε κατά πρώτο λόγο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον σε κάθε ε, θέμα εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ακολουθούν οι αγορητές εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Σάλβα. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Υπατή Εκπρόσωπη, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι θεωρούμε ότι η Λιτωνική Αμερική είναι ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, μια συμφωνία που αφορά 27 εκατομμύρια ανθρώπου και θα είναι η πιο φιλόδοξη περιφερειακή συμφωνία ανά τον κόσμο. Πιστεύουμε επίση ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική πριν από τη Σύνοδο τη Μαδρίτη που θα γίνει το Μάιο. Πιστεύουμε ακράδαντα στι συμφωνίε διασύνδεση με το Μεξικό και τη Χιλή, οι οποίε ήταν πραγματική επιτυχία και θα πρέπει να εκφράσουμε και την ικανοποίησή μα για τη σύναψη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κολομβία, η οποία θα είναι ευεργετική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη Λατινοαμερική αυτή χώρα. Θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κυρώσει αυτές τις ε, συμφωνίες ε, το συντομότερο δυνατόν και να διασφαλίσει ότι καμία από τις χώρες της κοινότητας των Άνδεων δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τις συμφωνίες. Οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μπορούν και θα πρέπει να είναι ένα χρήσιμο μέσο προκειμένου να ευνοείται η ανάπτυξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Τέλος, πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει αφενός να εμβαθύνουμε τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λοιπές χώρες, καθώς επίσης και να ευνοήσουμε και τις συμφωνίες ενδοπεριφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για την Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μενέντε Τεβάγε. Τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Άστον, Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συνάδελφο Σαλαφράγκα για την ε, θετική έκβαση της έκθεσής του. Γνωρίζετε ότι η Σύνοδος του Μαΐου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προαγάγουμε τις σχέσεις μεταξύ αμφωτέρων των πλευρών. Πρέπει να συγχαρούμε την Ισπανική Προεδρία για το έργο που επετέλεσε προς αυτόν τον στόχο. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι πρόκειται ε, ώστε σε σχέση με μετά την Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί αυτός ο συσχετισμός. Και εδώ πρέπει πολλά να γίνουν από πλευρά σας κυρία Άστον. <clears throat> Διότι σε σχέση με άλλη περιοχή που να έχει τέτοιες σχέσεις με την Ευρώπη, πολιτισμικές και ιστορικές, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περιοχή με τέτοιες σχέσεις. Και σε σχέση με την ίδια την βούληση των Λατινοαμερικανών, αλλά και σε σχέση με την βούληση των ε, Ευρωπαίων να υπάρξει υποστήριξη θεσμική, αυτό έχει πετύχει μια, ένα μεγάλο βαθμό παγίωση των σχέσεων. Αυτή η έκθεση που μπορούμε να πούμε ότι και η ομάδα μου συνεισέφερε θετικά υπέρ αυτής, είναι ένα θετικό μήνυμα για αυτή την Σύνοδο Κορυφή του Μαΐου στη Μαδρίτη και ελπίζω ότι θα μπορέσει να συνεισφέρει υπέρ των αποτελεσμάτων, θετικών αποτελεσμάτων αυτή τη Συνόδου. Και είναι επιτακτική ε, ε, ανάγκη να προχωρήσουμε στη στρατηγική διαμόρφωση αυτών των σχέσεών μα με τη Λατινική Αμερική και την περιοχή τη Καραϊβική. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα, στη δημιουργία ενός μηχανισμού επενδύσεων και στην ε, Eurolat. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι στη Μαδρίτη μπορεί να υπάρξει μια τελική προώθηση σε σχέση με την ολοκλήρωση της αγοράς αυτής. Ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Περού, την ε, Κολομβία και αναμένουμε ότι θα μπορέσει να εξευρεθεί μια διατύπωση ορθή και ευφυής που θα επιτρέπει τον επιθυμητό αυτό την, ε, την ένταξη, ευταία ένταξη του ε, η Περινού, του Εκουαδόρ και να υπάρξει και δυνατότητα που θα διανοείται για τη Βολιβία. Εν τέλει, πέρα από την ε, πιθανότητα θετική, πιθανότητα θετικής έκβασης ε, για τις διαπραγματεύσεις αυτές ε, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να δούμε και την προοπτική σε σχέση με τον Παναμά. Ολοκληρώνω Πρόεδρε λέγοντας ότι όλα αυτά πρέπει να βρουν απήχηση στο πλαίσιο που η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θεωρεί την κοινωνικο-οικονομική πολιτική που θα πρέπει να είναι το, τα βάθρα για μας. Υποστήριξη δηλαδή για την ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής, σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικέντρωση στα θέματα ανάπτυξης. Πάντα στοιχηματίζοντας στο διακύβευμα του να εξευρεθούν διάβλη διαλόγου και να εμβαθυνθεί έτσι η δυνατότητα της, ε, να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας ώστε να υπάρξουν πρόοδοι που θα σημειωθούν σε αυτούς τους τομείς. Σας ευχαριστώ. schön στα γερμανικά. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Στη συνέχεια ο κύριο Παναγιώτοφ για την Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στην Ευρώπη. Δύο λεπτά κύριε Παναγιώτοφ. Χωρίς μικρόφωνο. Microphone. Παρακαλώ με το μικρόφωνο τώρα. Okay. Σας ευχαριστώ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σαραφράγκα για την παρέμβασή του και τη συνεισφορά του για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τον ευχαριστώ και για την έκθεσή του. Η στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών της Λατινικής Αμερικής τα επόμενα χρόνια θα βρίσκεται ακριβώς στο πλαίσιο και στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη του 2020. Φυσικό είναι ότι θα λάβουμε υπόψη και θα προσέξουμε ιδιαίτερα και την οικονομία και το περιβάλλον μας. Τους στόχους ακριβώς για το περιβάλλον που πρέπει να είναι σεβαστή. Η Ευρώπη επλήγει με ιδιαίτερο τρόπο από την χρηματοοικονομική ε, κρίση και αυτή η εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Αμερικής διανοίγει νέες ευκαιρίες να μπορέσουμε να ε, ξεπεράσουμε αυτή την κρίση πιο γοργά και με καλύτερο τρόπο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λούνατσεκ τώρα για τους πράσινους και την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικό, τουλάχιστον για το. Θα μιλήσω στο πρώτο τμήμα μου ισπανικά. Θέλω και εγώ να αναγνωρίσω σε αυτή τη διαδικασία την ε, προώθηση που δόθηκε ε, σε σχέση με την παρουσίαση τη έκθεση ε, Σαλαφράγκα και αυτού που καταφέραμε μέχρι τώρα. Και είναι νομίζω θετικό αυτό, αυτό το οποίο πετύχαμε. Ένα τρόπο θετικό γιατί εσεί δεχθήκατε πολλέ δικέ μα προτάσει και θέσει. Και θα έπρεπε να πω ότι αν ήταν μια έκθεση των Πρασίνων θα ήταν ίσως διαφορετική όμως αυτό συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως θα ήθελα να πω σε σχέση με τον κύριο Σαλαφράγκα θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής ως σχέσεις μεταξύ ίσων. Θα μου άρεσε αυτή η ιδέα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν είναι ίση η σχέση αυτή. Έχουμε εδώ και τις κυβερνήσεις αλλά και τους φτωχούς ε, που ζητούν περισσότερα δικαιώματα και χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες όπως και οι γυναίκες ή και την καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καθορίσουμε περισσότερο. Είναι κάτι που βλέπω ότι απουσιάζει ακόμα από την έκθεση. Όμω έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου εξ ονόματο των Πρασίνων, διότι καταφέραμε τα δικαιώματα των αυτοχθόνων να τα εντάξουμε σε σχέση και με τι δυνατότητε για την ανάπτυξη και την, ε, τις πολιτισμικές ε, ε, πτυχές και σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες επίσης τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεγάλε πρόοδοι αυτές για τις κλιματικές αλλαγές ε, που έχει εξίσου επιπτώσεις ε, στους ε, ανθρώπους αυτής της Υπήρου. Για παράδειγμα στο τι συμβαίνει με την τήξη των παγετώνων εδώ υπάρχουν ακόμα και διαφορές μεταξύ αυτών που εμείς θα θέλαμε να μπορέσουμε να περάσουμε οι πράσινοι ε, και ε, άλλοι. Δεν είμαστε υπέρ του να συνεχιστούν ε, οι συμφωνίες εταιρική σχέσης όπως έγινε. Η κοινότητα των Άνδεων θα έπρεπε σε σχέση με τις χώρες των, της κοινότητας των Άνδεων θα έπρεπε να έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία και όχι μόνο με κάποιες ξεχωριστές χώρες όπως την Κολομβία ή το Περού. Θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά είναι μια ερώτηση, ένα θέμα που τίθεται προς εμά, είπατε εκπρόσωπε, ε, αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να εντάξουμε στην έκθεση δυστυχώς. Και αυτό είναι το να είμαστε κατά των τεράστιων αυτών ε, προγραμμάτων, τεχνικών, τεχνολογικών προγραμμάτων όπως ε, το φράγμα στο, ποτάμι, στο ποταμό Σιγκού και που καταστρέφει την περιοχή των ε, Ιθαγενών ε, Ινδιάνων. Υπάρχει εδώ και ακριβώς στην, στην ίδια τη Βραζιλία το θέμα των πολλών οργανώσεων που δίνουν μάχη κατά αυτού του εγχειρήματος. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς ως είπατε εκπρόσωπος, τι κάνετε σε σχέση με την προστασία της περιοχής του Αμαζονίου και την προστασία των ηθαγενών που ζουν στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Ήμουν πραγματικά γενναιόδοροι απέναντί σα, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Στην συνέχεια για του Ευρωπαίους συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριος Τάνοκ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Συγχαίρω τον Νάτσο Σαλαφράγκα για μια εξαιρετική έκθεση όσον αφορά τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική. Μετά τη διεύρυνση του 2004 με τι χώρε τη Κεντροανατολική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικέντρωσε και είναι κατανοητό αυτό στι σχέσει τη προ την Ανατολή σε σχέση με αυτέ τι χώρε, τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, οι, σχέσεις, οι εμπορικέ μα σχέσει με τι χώρε τη ε, ε, αναπτύσσονται ταχαίω. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτέ τι χώρε η Βραζιλία ε, και άλλες χώρες, αναδυόμενες χώρες ε, ε, και σε σχέση με την, τις εκλογές όταν ο πρόεδρος Λούλαντα Σίλβα αποχωρήσει η Βραζιλία και το Μεξικό καθορίζονται ως στρατηγική σημασία σε τέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κολομβία πολλά υπόσχεται για το πώς μπορεί μια δημοκρατία να ανθίσει στη Λατινική Αμερική και διαπραγματεύεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κολομβία. Θα γίνουν προεδρικές εκλογές και εκεί. Και εδώ σε σχέση με τον ηγετικό ρόλο του Άλβαρο Ουρίμπε είναι πολλοί οι οποίοι ε, θα ήθελαν να υπάρξει συνέχεια. Εδώ σε σχέση με τη δημοκρατία και την ελευθερία της, έκφραση. έκφρασης η Βολιβία και ο Ισημερινός έχουν ε, δώσει ανησυχητικά μηνύματα σε σχέση με τα όσα κάνει ο πρόεδρος Τσάβε στη Βενεζουέλα και στα όσα συμβαίνουν στην Κούβα από πλευρά του κυρίου Κάστρο. Εδώ σε σχέση με άλλες χώρες ε, για παράδειγμα ε, γίνεται ε, χρήση σε σχέση με την Αργεντινή ενός ε, λεξιλόγιου που θυμίζει πολεμικό, πολεμική ορολογία όσον αφορά την Μεγάλη Βρετανία και τα νησιά Μαλβίνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια Μπέντερ, μισή λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω ότι η έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λατινική Αμερική. Με, κάνει, με ε, ικανοποιεί ιδιαίτερα για το ότι είναι παρούσα η κυρία Άστον. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι το σύνολο της Νότιας Αμερικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η Βραζιλία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, επίλυση σε σχέση με το πυρηνικό πρόβλημα που υπάρχει με το Ιράν. τα στενότερη συνεργασία με την Λατινική Αμερική όσον αφορά την καταπολέμηση των ε, Ισλαμικών δικτύων τρομοκρατών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ε, Βενεζουέλα. Ένα τρίτο σημείο, στενότερη συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής όσον αφορά την παγκόσμια καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές ανησυχίες μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Τσάβες στη Βενεζουέλα, αλλά όχι μόνο αυτού. Πρόσφατα είχαμε μία έκθεση όσον αφορά την κατάσταση στην Λατινική Αμερική και στον τύπο ε, αναφέρεται η προέλαση της Κίνας σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ πώς θα μπορούσαμε να καθορίσουμε τον ρόλο των στρατηγικών εταίρων. Για τους μη εγγεγραμμένους 1,5 λεπτό κύριος Γκόλνης παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα έχει συμπεριλάβει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι πληρέστατη, δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται η σχέση, για τη σχέση της Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, ε χώρες ε, που ε, αντιστοιχούν ε, σε 600 εκατομμύρια άτομα, 10% ε, του παγκοσμίου ΑΕΠ και με τους οποίους έχουμε ένα παρελθόν ιστορικό, ειδικότερα όσον αφορά την Ισπανία, την Πορτογαλία και η Ιταλία που πάρα πολλοί Ιταλοί πήγαν στην Αργεντινή. Και αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι δεν αναφέρεται σε δύο ε, ζητήματα πολύ σημαντικά. Το θέμα των ελεύθερων ε, συναλλαγών ε, με την περιοχή αυτή, όπως επίσης τις συνθήκες εργασίας και τα σχετικά ζητήματα που παρουσιάζονται ως πανάκια γενικότερα και που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική την ίδια. Δεύτερον, το πρόβλημα της ανεξαρτησίας σε σχέση με τον με τον μεγάλο αδερφό, τον Big Brother, ε, τους Αμερικανούς. Εμείς δεν είμαστε κακοί. Το δόγμα Μονρόε που είχε σκοπό τότε να μην υπάρξει επαναπικιοποίηση ε, της ε, Λατινικής Αμερικής από την Ευρώπη έγινε προτεκτοράτο τελικά γιατί πριν από μερικά χρόνια είδαμε τα αποτελέσματα όλης αυτής της δυνατότητας, όλης αυτής της κατάστασης μέσω της κατάστασης που πήγε στον Παναμά. Ε, όσον αφορά τώρα τα ε, ναρκωτικά, δεν μπορούμε να πούμε στους ε, πολίτες Λατινικής Αμερικής να αναφερθούμε μόνο στα ζητήματα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Πρέπει να επικεντρωθούμε και σε άλλα ζητήματα που είναι εξίσου σημαντικά. Ακολουθούν οι άλλοι αγορητές σε αυτή τη συζήτηση. Μπασέσκου, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι. Κυρίως θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σαλαφράγκα για την εξαιρετική του αυτή έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβιβάζει αυτή τη στιγμή ένα σαφές μήνυμα εντατοποίηση των σχέσεων με τη, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Μια και μέσα ένα μήνα θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, αυτή η Ένωση ε, είναι αυτή η σχέση είναι μια προτεραιότητα επίσης και της Ισπανικής Προεδρίας. Πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό το οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε για να αυξήσουμε τις συναλλαγές μας μεταξύ αυτών των δύο περιφερειών χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα κονδύλια ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να προαγάγουμε τις, ε, τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στι ε, αγορέ Λατινική Αμερική. Υπάρχουν προϊόντα τη Ρουμανία που έχουν και θέση εκεί, όπω και το προϊόν μα τη αυτοκινητοβιομηχανία μα τη Ρουμανία, το αυτοκίνητο Ντάτσα στη Λατινική Αμερική. Έχουμε λοιπόν μέσα στο πλαίσιο αυτή τη εταιρική σχέση κοινέ αξίε και είναι λοιπόν ε, ευπρόσδεκτα αυτά τα οποία προτείνονται. Πρέπει να αποτελέσουν μέρο ε, των σχέσεων τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με την Λατινική Αμερική. Είδαμε επίση προγράμματα που θα παγιώνουν το νομικό καθεστώ των γυναικών ένα, σε ένα ισότιμο πλαίσιο για την απασχόληση, την παιδεία και την απασχόληση. Ολοκληρώνω η έκθεση αυτή Σαλαφράγκα σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατίνική Αμερική πρέπει να είναι τα βάθρα, η βάση αυτών των σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος ε, Χαουρέγγι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου σα συγχαρητήρια προ τον κύριο Σαλαφράγκα. Είναι μια έκθεση πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας πω κύριε και κύριοι ότι υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι για να θεωρούμε τη Λατινική Αμερική ω μια πολύ σημαντική ήπειρο για την Ευρώπη. Υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν στη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν εκατομμύρια Λατινοαμερικανών που ήρθαν στη χώρα μα, ήρθαν στην Ισπανία, ήρθαν στην Ευρώπη, που βρήκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Ισπανία χώρε υποδοχή, χώρε ασύλου για τα δεινά, τα πάνδυνα που περνούσαν στη Λατινική Αμερική αυτή η λαοί. Είναι πάρα πολύ σημαντική κυρίε και κύριοι η Λατινική Αμερική για την Ευρώπη. Γι' αυτό χαίρομαι, εκφράζω την ικανοποίησή μου ότι του επόμενου μήνε, ίσω σαν συνέπεια τη εργασία ε, τη κυρία Άστον και τη Ισπανική Προεδρία, θα είναι δυνατόν να υπάρξουν τέσσερι συμφωνίε πολύ σημαντικέ με την Κολομβία, με το Περού, να ξεκινήσει και με το Μερκοσούρ συμφωνίε ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω και για τη Λατινική Αμερική. Η Λατινική Αμερική Αμερική είναι κάτι που πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι κράτη ευάλωτα, ε, Είναι ε, δημόσιες υπηρεσίες πολύ ευάλωτες και πρέπει να βοηθηθούν. Έχουν δημοκρατίες που είναι στα σπάργανα ακόμα και έχουν ατέλειες. Υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι αυτές τις χώρες. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη σχέση και αυτή την προοπτική, αυτό το όραμα. Θέλω να δώσω δύο μηνύματα, δύο συστάσεις κυρία Άστον, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Για να δουλέψουμε στη Λατινική Αμερική πρέπει να βασιζόμαστε επίση και στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Η εξωτερική μα πολιτική, κύριε Άστον, πρέπει να γίνεται με μια πολύ ισχυρή οικονομική παρουσία δική μα μέσω αυτών των εταιριών στη Λατινική Αμερική, που μπορούν πάρα πολύ να συνεισφέρουν για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Με, μια, με ένα πολιτισμό κοινωνική υπευθυνότητα και ευθύνη σε αυτέ τι χώρε και δέσμευση υπέρ τη ανάπτυξη αυτών των χωρών. Και τέλο, πρέπει να έχουμε μια γενική ε, συμμαχία με τη Λατινική Αμερική, να είμαστε σύμμαχοι για να συνεργαστούμε για τη διακυβέρνηση του κόσμου και να είμαστε πιο ισχυροί. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο η κυρία Μάισνερ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Άστον και αγαπητέ κύριε Σαλαφράγκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την έκθεσή σα ε, ως μέλος της ε, ομάδας Ευρωλάτ, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής να εντείνονται και να ενδυναμώνονται διαρκώ. Από το 1999 πολλέ προόδου έχουμε σημειώσει. 600 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη Λατινική Αμερική <clears throat> περίπου 600 εκατομμύρια στην ε, Ευρώπη. Και έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες. Η επιθυμία για την ειρήνη και τη δημοκρατία μας ενώνουν. Όμως οι όροι και προϋποθέσεις είναι διαφορετικοί πάντα. Οι εταίροι πρέπει να προσέχουν να είναι εξίσου ισχυροί. Δεν είμαστε όμως εξίσου ισχυροί ακόμα οι Λατινοαμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Έχει πολλά προβλήματα με τον αναλφαβητισμό, αναλφαβητισμό η Λατινική Αμερική, με ελλειπείς υποδομές, με προβλήματα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ε, δεν έχουμε σε αυτό το τομέα τόσα προβλήματα. Έχουμε όμω προβλήματα με τα ναρκωτικά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ω εταίροι. Είναι δουλειά μα ω σημαντική εμπορική εταίρη και για την ανάπτυξη όσον αφορά το εμπόριο σε σχέση με τι χώρε τη Λατινική Αμερική να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ στον εκδημοκρατισμό του. Θα έλπιζα η εταιρική σχέση να οδηγήσει ώστε η Λατινική Αμερική να μπορούν να ζουν σε ένα καθεστώ ειρήνη οι πολίτε οι άνθρωποι όπω ζούμε και εμεί σε ένα καθεστώ Ειρηνή εν ειρήνη στην Ευρώπη και να μπορούν να μάθουν ένα από τον άλλο. Και γι' αυτό μου αρέσει η ιδέα της ε, ε, ευρω... λατινικής, λατινοαμερικανικής ε, εταιρικής σχέσης υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας. Νομίζω αυτό θα εμβάθυνε ακόμα περισσότερο την εταιρική μας σχέση και θα ήταν πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Κουσούφνικ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, Ο συνάδελφος Αλαφράνκα ανέφερε στην αρχή ότι οι αρχές μας είναι παρόμοιες με αυτές της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχει όμως και ένα αλλά και το συζητήσαμε στο πλαίσιο της ε, συνόδου με τη Λατινική Αμερική. Το θέμα της Κούβας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κούβα έξω. Ε, από το πλαίσιο αυτό. Όμω, λόγω του καθεστώτο τη Κούβα, δημιουργούνται πολλά προβλήματα για ολόκληρη την περιφέρεια. Η περιφέρεια όμω ε, υποφέρει από αυτό. Είναι σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο εταίρο μα δεν μπορεί να είναι το καθεστώς του Κάστρο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το καθεστώ του Κάστρο και θα ήθελα τον Καρδινάλιο Γαρίο Ορτέκα να τον ε, ε, ευχαριστήσω για τι προσπάθειε που έκανε όσον αφορά την ενίσχυση του κράτου δικαίου, το σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί αυτό είναι μια βάση και απαραίτητη, προ... Ε, προπόθεση για την δημοκρατία. κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή της συζήτησης η Βαρόνι Άστον είπε ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ε, ευγένεια της, σας ζητώ κυρία Άστον να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνει και τις διαπραγματεύσεις για, την, για τον καθορισμό μιας ε, χάρτας που θα βασίζεται στη Χάρτα των Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ποιανόν τα συμφέροντα ε, εξυπηρετούνται στην Αργεντινή όταν ζητήθηκε ε, ε, επισήμω από τα Ηνωμένα Όθηνα να βοηθήσουν να σταματήσουν οι μονομερές πράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, εξόριξη πετρελαίου στην περιοχή. Οι Λατινοαμερικάνοι ηγέτες στήριξαν ομόφωνα την απόφαση αυτή και το αίτημα της Αργεντινής. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών ε, δίνει δικαίωμα στη Βρετανία να υποστηρίζει τα δικαιώματα αυτά. Εσείς ποιον θα υποστηρίξετε σε αυτή τη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. κυρία Βέρτμαν, ένα λεπτό παρακαλώ. Επόμενη. Αγαπητοί συνάδελφοι, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής υφίσταται από το 1999 μια διμερής στρατηγική εταιρική σχέση. Ένα πυλώνα θεμελιώδη αυτή τη εταιρική σχέση είναι ο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό ο πυλώνα, ωστόσο, παραβιάζεται πολύ συχνά και βλέπουμε ότι σε σχέση με πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους στη Λατινική Αμερική είναι ακόμα αναλφάβητοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα σημαντικό εταίρος ε, της, ε, των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Κοινωνικά είναι σε μειονεκτική θέση οι γυναίκες ε, και ασκούν αρνητικές διακριτικές μεταχειρήσεις εις βάρος τους. Και όλα αυτά βρίσκονται σε αντίφαση με τα ενισχύ ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Επόμενη η κυρία Γιαννάκου, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κύριο Σαλαφράνκα για την ιδιαίτερα ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεσή του και θέλω να συμφωνήσω επίσης με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, για τη σημασία που δίνει στην προσπάθεια αυτή για μια εταιρική σχέση πολύ πιο στενά συνδεδεμένη είναι γεγονό ότι στη λατινική αμερική έχουν υπάρξει εξελίξει κατά την τελευταία εικοσαετία και είναι αλήθεια ότι αυτά που μα απασχολούσαν κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1980, δηλαδή πολλέ δικτατορίε, έχουν εξαλειφθεί. Ωστόσο δεν έχει εξαλειφθεί το εμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα μαύρου χρήματο, η τρομοκρατία και τα μεγάλα προβλήματα που προέρχονται από τη φτώχεια, την ανασφάλεια και την ανεργία στην περιοχή. Καλούμε με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Βαρόνια Άστον να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε τομείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. οι χώρες της λατινικής αμερικής είναι οι μόνες χώρες που μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται τόσο στενά από οποιασδήποτε τρίτες χώρες με την ευρώπη σε θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία με την παιδεία έχουν σχέση με τον πολιτισμό και νομίζω ότι σε αυτούς τους τομείς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. η έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προτείνει άλλωστε τη δημιουργία ενός ιδρύματος που έχει τεράστια σημασία και για το ευρωκοινοβούλιο και βεβαίω ζητεί ένα καινούριο ρόλο και πιο ισχυρό για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στη σχέση με τις χώρες αυτές και νομίζω κυρία πρόεδρε ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή έκθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μποσκούρτ, δύο λεπτά, επόμενη αγορήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες η Λατινική Αμερική όλο και πιο συγκεκριμένα βρισκόταν στο επίκεντρο της προσοχής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δεκαετίες ε, που είχαμε παραμελήσει τις χώρες ε, της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στρατηγική εταιρική σχέση με σημαντικούς εταίρους στρατηγικής σημασίας χώρες δηλαδή της Νότιας Αμερικής. Εδώ πρέπει να δούμε επίσης και την, τις συμφωνίες σύνδεση με χώρε της Κεντρικής Αμερικής. Βρισκόμαστε στο τελευταίο γύρο, έχουν, έχουμε διαπραγματευτεί ε, πολλά θέματα, απομένουν λεπτομέρειες, θα ολοκληρωθούν αυτές οι συμφωνίες. Χαιρετίζουμε τις συμφωνίες με τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής, όμως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογραμμίζω ότι πρέπει να έχει πριτανεύοντα ρόλο. Θα πρέπει η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Αμερική να βελτιωθεί και να δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε αυτές οι χώρες ε, πραγματικά να σέβονται και να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επομίζεται ιδιαίτερες ευθύνες ε, ακόμα και μετά την ε, σύναψη αυτών των ε, συμφωνιών. Δεν πρόκειται μόνο για αυτές τις συμφωνίες, για πολιτικό διάλογο και συνεργασία. Η Συμφωνία Σύνδεσης για τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής έχει τεράστια σημασία. Αυτή η περιοχή του κόσμου πλήττεται από τη φτώχεια και πρέπει να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε υπέρ της ανάπτυξης των χωρών αυτής της περιφέρειας. Στις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ότι τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισότιμοι εταίροι μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής σχέσης, διότι είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση μεταξύ τους. Είναι μια ασυμμετρική θα έλεγα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών αυτών. Πρέπει να μεριμνήσουμε λοιπόν όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκομίζουν τα κέρδη από αυτή την ε, εταιρική σχέση, αλλά κυρίως η ζωή των πολιτών να βελτιωθεί. Έχουμε επιλέξει αυτή την πορεία και θέλω να τονίσω ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν και όλες οι χώρες της περιοχής αυτής να συμπεριληφθούν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ο επόμενος αγορητής Airworld, ένα λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο θέμα του εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Λατινικής Εμορικής. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο γίνεται ε, σε ένα ισότιμο πεδίο καλλιεργητέ και παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαίνονται πολλού κανόνε και παράγουν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Αυτέ οι υψηλέ προδιαγραφέ ε, σημαίνει ότι έχουμε και επιπλέον κόστο για την παραγωγή για του καλλιεργητέ ε, στην Ευρώπη και επομένω μπορεί να βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα και αγαθά που είναι κατώτερη ποιότητα και παράγονται με κατώτερο κόστο. Και αυτά δεν είναι μόνο προ όφελο των Ευρωπαίων παραγωγών. Δεν θα πρέπει να το σκεφτούμε μόνο προ όφελό του, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για την ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρώπη δεν ε, παραβιάζουν συγκεκριμένου κανόνε και δεν διακυβεύεται η υγεία των καταναλωτών με τη χρήση του και την κατανάλωσή του. ξεπεράσατε τον χρόνο σας κατά πολύ. Είχατε ένα λεπτό. Θέλετε να ολοκληρώσετε ίσως την πρότασή σας αυτή. Υπάρχουν 600 εκατομμύρια κάτοικοι στη Λατινική Αμερική και το ΑΕΠ τους είναι το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και η δυνατότητα ενίσχυσης των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκμεταλλευτούμε αυτή τη ε, δυνατότητα. Πολύ ωραία μεγάλη πρόταση αυτή που εκφωνήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιγκάτσκι παρακαλώ και αυτό σε ένα λεπτό τώρα επόμενος. Σας ευχαριστώ θα προσπαθήσω πραγματικά να τηρήσω αυτό το χρονικό όριο του, λεπ, του ενός λεπτού. Κυρίε και κύριοι, ο Φουκουγιάμα δεν είχε μάλλον δίκιο όταν είπε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία ήταν το τέλος της ιστορίας. Σίγουρα όμως είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η, ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό καθεστώς είναι το καλύτερο μέσα στο οποίο μπορούν να ζουν ε, οι άνθρωποι. Δυστυχώς όμως αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική είναι το αντίθετο. Έχουμε εδώ ένα αντικατάσταση της ε, δημοκρατίας από ε, λαϊκιστικό, σοσιαλιστικό καθεστώ. Γι' αυτό απευθύνομαι προ την ε, κυρία Άστον. Και θα ήθελα να πω ότι η δική μας πείρα και στα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και η δική μας τεχνογνωσία πρέπει να περνάνε σε χώρες ε, με, ε, όχι σε, ε, με δικτατορικό καθεστώς αλλά σε δημοκρατικές χώρες. Σας ευχαριστώ. Θα λάβει τον λόγο στη συνέχεια Κρέτου 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, οι σχέσεις με τη Λατινική Αμερική έχουν τη σημασία τους από την πρώτη στιγμή μέχρι τη στιγμή ανάπτυξης αυτών των σχέσεων. Αυτή η στρατηγική σχέση έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις σχέσεις μας ε, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για πάνω από τρία δις ε, τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, μέχρι σήμερα, οι χώρες αυτές μπόρεσαν να αντέξουν τη χρηματοοικονομική κρίση με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ότι αναπτυγμένα κράτη. Έχουμε βέβαια και ένα ε, επίπεδο φτώχεια. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν, μαστίζονται από χρόνια προβλήματα και από τα προβλήματα της κακοδιαχείρισης. Ε, στη Βολιβία μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Σε άλλες χώρες το επίπεδο είναι ανώτερο. Για παράδειγμα στην ε, Αργεντινή το 13,9 ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Γι' αυτό η υποστήριξη για την ανάπτυξη πρέπει να επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του θεσμικού δυναμικού αυτών των χωρών και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να απαμβλύνουμε τις ε, ε, οξύες αυτές ε, αντιθέσεις. Πρέπει να υπάρξει διάλογος, να προωθήσουμε τον διάλογο για να υλοποιήσουμε τους στόχους της ανάπτυξης της χιλιετίας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η στρατηγική θα συμπεριλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις ΜΚΟ που θα πρέπει να συμμετέχουν συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο για την ανάπτυξη αυτών των στόχων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, Μακλάρκιν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω μέλο τη Eurolat, θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία και τον κύριο Σαλαφρέγκα, ο οποίο επεσήμανε τη σημασία των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική. Η αλλαγή του κλίματο θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τι χώρε τη Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική και οι στόχοι ε, για τη μείωση των εκπομπών θα πρέπει να ενισχυθούν. Τέλο, ε, επιπλέον, συγγνώμη, ο διάλογο για την ενέργεια θα πρέπει ε, να συνεχιστεί και θα πρέπει να συνδράμουμε για να έχουμε βιώσιμη κατανάλωση ενέργεια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη παιδεία και ο τελικό στόχο μα θα είναι οι σχέσει μα με τη Λατινική Αμερική να αποτελέσουν ε, το ένασμα για βελτιωμένη παιδεία και θα πρέπει επίση να βελτιώσουμε την ε, προαγωγή του εράσμου στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τι εξαιρετικέ δυνατότητε που μπορούν να προσφέρουν ε, για την επαγγελματική ανέλυξη και για τις τη μελλοντική σύσφυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωση Λατινική Λατινικής Ευχαριστώ. Είμαστε στο τέλος ε, της συζήτησης. Περνάμε στο Catch the Eye. Πρώτος ο κύριος Νικολάζητς για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, καλωσορίζω την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής που είναι βεβαίως στόχος ε, και της Ισπανικής Προεδρίας και αμοιβαία επωφελής και μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Η Λατινική Αμερική έχει τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, πάνω από 600 εκατομμύρια κατοίκους. Βεβαίως και η φυσική της ε, πόρη είναι πλούσιοι και έχει ένα ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ που φτάνει το 10%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος Λατινικής Αμερικής και πρέπει να εδραιώσει την θέση της. Η πλήρως λειτουργική συνεργασία που βασίζεται σε κοινέ αξίε όπω η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα απαιτήσει στοχευμένη βελτίωση τη ε, περιφερειακής μας σχέσης. Ε, εγώ θα υποστηρίξω τα ίδια και στην Γιούρλαντ στην Ισπανία στη δεύτερη διάσκεψη. Ευχαριστώ επόμενη συνάδελφη η επόμενη συνάδελφη μας την κυρία Κρίσμπεκ αλλά δεν είναι στην αίθουσα έφυγε οπότε περνάμε στον κύριο Ρωμέβα συγγνώμη για τα ισπανικά μου ο κύριος Ρωμέβα για ένα λεπτό Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία προκειμένου να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ζήτημα. Η κατάσταση που γνωρίσαμε πριν από μερικέ μέρε και που έχει σχέση με την Κολομβία. Ανακαλύφθηκε η άμεση ε, εμπλοκή, των, ε, των δυνάμεων ασφαλείας σε ό,τι φορά την δίωξη και την ε, δημιουργία κάποιων ψευδομαρτύρων προκειμένου να ε, κατηγορήσουν ε, κάποια άτομα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ ανησυχητικό. Σε αυτή την ε, πληροφορία που έλαβα έμαθα ότι από πλευράς κυβέρνησης της Κολομβίας φροντίζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευδείς σχέσεις με τους ΦΑΡΚ και πέραν αυτού αυτό που είπε η κυρία Φάρκ για την ευρωπαϊκή συνεργασία νομίζουμε ότι αυτό δεν έχει αποβεί σε όφελος της συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απαιτεί ε, συζήτηση με την κολομβιανή κυβέρνηση και χρειάζεται η κολομβιανή κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έπραξε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μόλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από 300 χρόνια επικαιοκρατίας και μετά από τον ψυχρό πόλεμο η Λατινική Αμερική αναπτύσσεται το ότι ο πρόεδρος ε, της Ρωσίας Μετβέντεφ ταξίδεψε ως εκεί αποδεικνύει πως προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις του με την Νότια Αμερική και το πόσο σωστή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη σημασία που αποδίδει σε μια περιοχή που έχει περισσότερους κατοίκους από την Ένωση των 27. Βεβαίω αυτό δεν αφορά μόνο το Μερκοσούρα, αλλά να σκεφτούμε και τι μικρές χώρε που δεν ανήκουν σε αυτή την κοινότητα ή στην κοινότητα των Άνδεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο κύριος επενδυτής και δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. Από οικονομική πλευρά νομίζω είμαστε σημαντικότεροι και πρέπει να καταληθούμε αυτή την pole position που έχουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Μόλτσερ. Τον λόγο έχει ο κύριος Σιλβέστρης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική έχουν αναπτύξει μια στρατηγική συμμαχία, ε, εταιρική σχέση γνώμη, προκειμένου να ε, βελτιωθεί η ανάπτυξη τη περιοχή αυτή. Από το 1999 συνεχίζουν οι διμερεί συνεργασίε και οι διμερεί συναντήσει. Η προσοχή θα έρθει στη Μαδρίτη το Μάιο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λαμβάνω το λόγο σήμερα και ε, θα ήθελα να υπερασπιστώ την έκθεση του συνέλφου Σαλαφράγκα. Θα ήθελα και εγώ, όπω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, συνεχάρισαν τον εισηγητή. Είναι κάτι το δικαιολογημένο. Η έκθεση στοχεύει στο να ενισχύσει περαιτέρω τι σχέσει που υπάρχουν ανάμεσα στι δύο περιοχέ σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Και έτσι η πρωτοβουλία ε, για τη σύσταση ενό ιδρύματο είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο επίκαιρο. Μέλο τη Επιτροπή Γεωργία, θα ήθελα να τονίσω αυτή την τελευταία πτυχή τη οικονομία, αναφέροντα κάποια στοιχεία για να καταδείξω ότι πρόκειται για μια ζώνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί κατοικούν 600 εκατομμύρια πολίτε και παράγουν πολλέ πρώτε ύλε. Τελευταία επηρεάστηκε η γεωργική παραγωγή από τις καιρικέ συνθήκες θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτο επενδυτή στην Λατινική Αμερική και ο πρώτο δωρητή και έχει, ε, ε, έχει επενδύσει 30 ε, δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στη σημασία που έχουν οι σχέσει μας και ό,τι αφορά τη δημιουργία περαιτέρω διαλόγου για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και την επίτευξη των στόχων τη Κοπεχάγη. Σε συνεργασία με τι αναπτυσσόμενε χώρε, ε, αυτό είναι ιδιαίτερα ουσιώδε για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει εμεί ω Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιλβέστρη. Ο κύριο Καζίνη έχει το λόγο. Απουσιάζει. Ο κύριος Σκίν. Παρακαλώ. πω. Πώς θέλω να σας συγχαρώ για όσα έγιναν και για τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Αλλά όπως κάποιοι επισημάνουν, πα, επισημαίνουν, παραμένουν κάποια δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την Κολομβία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν συναδελφών όπως ο Ρίτσαρτ Χάουιτ που λείπει λόγω ηφαιστείων όπως ξέρετε, πρέπει να πούμε πως έχει επισημάνει ιδιαίτερα τα προβλήματα των συνδικαλιστών στην Κολομβία και θέλω να ζητήσω από την Επίτροπο να το λάβει αυτό υπόψη σε οποιαδήποτε στρατηγική και εμπλοκή έχουμε εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τον λόγο έχει η κυρία Άστον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να ξεκινήσω και εγώ όπως και οι κυρίες και κύριοι βουλευτές συγχαίροντας τον κύριο Σαλαφράγκα για την έκθεσή του και την Ισπανική Προεδρία για το έργο το οποίο έχει κάνει όχι μόνο προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής αλλά στηρίζοντας και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί είναι σημαντική η Σύνοδος, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την σχέση την οποία ανέφεραν οι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα έχουμε και μία Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών που για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο σημαντικό για να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να εμβαθυνθεί η σχέση με διάφορα παρόντα κράτη. Επίσης μιλήσαμε για τη σημασία του εμπορίου και τον ρόλο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είμαστε ο μεγαλύτερο επενδυτής στην περιοχή και χαίρομαι που οι συνάδελφοι ανέφεραν τον ρόλο της καινοτομία, που είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, μεγάλη έμφαση και στα ανθρώπινα δικαιώματα η σημασία του να διασφαλίσουμε πως αποτελούν κομμάτι της δυναμικής σχέσης που έχουμε και συμπεριλαμβάνει όλοι μας όλη μας τη δουλειά. Επίσης αναφέρατε την πλευρά του φεμινισμού των αυτοχθόνων λαών που πάντα οι Κομισιόν τις υπερασπίζονταν και ιδιαίτερα γνωρίζω τις απόψεις που επικρατούν και εδώ μέσα βεβαίως στην διεθνή ε, κοινότητα συνεχίζουμε λοιπόν να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σημειώνουμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί και οι συνάδελφοι θα δουν πράγματι τι σημασία έχουν οι ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εμπορική αυτή συμφωνία καθώς νομίζω πως ε, θα προχωρήσουμε αρκετά για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των συναδέλφων όσον αφορά την Κολομβία. Συμφωνώ επίσης για το ρόλο που παίζουν αυτές οι χώρες ε, στις γενικότερες διεθνείς σχέσεις αναφέρθηκε η Βραζιλία σε σχέση με το Ιράν. Είχα έρθει επαφή με τον Πρωθυπουργό της ε, Βραζιλίας ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Τα νησιά Φόρκλαντ αναφέρθηκαν βεβαίως στα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσση. πρόκειται λοιπόν για μια συνδεδεμένη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει να ισχύσει το κράτος δικαίου κλιματική αλλαγή και εκεί πέρα υπάρχει διάλογος κλειδί και βεβαίως χάρηκα ιδιαίτερα για το ότι αναφέρθηκε και το εράσμος. Και πάλι λοιπόν ευχαριστώ τον κύριο Σαλαφράγκα. Thank you very much, Mrs. Ashton. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άστον. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να πω κύριε Άστον πως το βασικό στοιχείο ε, το οποίο βασίζεται η έκθεση αυτή για τα προσοχή έτη είναι η κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης. Υπήρχαν πολιτικές λόγοι για τους οποίους προχώρησαμε στο 1985 στο διάλογο του Σαν Χωσέ και ήταν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους προχωρήσαμε στην θεσμοθέτηση του διαλόγου το 1990 και ήταν πολιτική λόγοι για τη συνέχιση αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να πω στου αδέλφου ότι πράγματι είμαστε μια κοινωνία αξιών και να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια εγκρίναμε ένα σημαντικό ψηφίσμα για την Κούβα όπου ζητάμε την άμεση απελευθέρωση και άνευ όρων των πολιτικών κρατουμένων. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Άστον προκειμένου να ενεργήσει έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο Ιντραρόκε, ο οποίος απόκτησε την Ισπανική ε, ηθαγένεια αλλά και του Φερνάντο Φερνάνδε Μαρτίν για να μπορέσει να ε, μεταβεί στην Ισπανία. Θα ήθελα να πω Τώρα, να περάσουμε δηλαδή από τα λόγια στην πράξη και αναφέρουμε στην Συμφωνία Σύνδεση. Κυρία Άστον, εσεί διαπραγματευτείτε πολύ σωστά τη Συμφωνία τη Κολομβία και του Περού. Αλλά πιστεύω πω η κατάσταση πρώτον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και είναι ανησυχητική στην Κολομβία, ε, βελτιώθηκε σημαντικά και νομίζω ότι ο λαό τη ε, Κολομβίας αξίζει να ζήσει μέσα σε ειρήνη. Πιστεύω ότι και η πλησφέρεια του Κοινοβουλίου συμφωνεί με αυτήν τη ε, συμφωνία. Ε, θα ήθελα κυρία Άστον να πω ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο οξυγόνο στο πλαίσιο των διαπραγματευτών Εμεί αποτελούμε το 25% των εξαγωγών του και αυτοί αποτελούν το 2% των δικών μα. Θα πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι και να προωθήσουμε τη συνεργασία με το Μερκοσούρ. Νομίζω κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω, πω η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κατάσταση παρακμής από οικονομικής σκοπιάς. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προσδοκούμε από την υπάτη ε, εκπρόσωπο να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάσκεψη της Μαδρίτης και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο της ε, Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με Ελληνική Μερική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η εξουφορία θα διεξαχθεί στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Σε ό,τι αφορά την μίληση διάταξη της ε, αυριανής